Buon pomeriggio e benvenuto a tutti. Καλό από μεσήμερο και καλώ ήρθατε όλε και όλοι. Se vi accomodate possiamo cominciare. Όταν καθίσετε θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Oggi pomeriggio tocca a me presiedere. Σήμερα ο κλήρος πέθησε μένα προκειμένου να προεδρεύσω στη συνεδρίαση της Επιτροπής διότι είμαι ο μοναδικός επιζήσας από την προηγούμενη θητεία. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης και σας υπενθυμίσω πως η μέσα διάταξη της σήμερα είναι η εξής. θα πρέπει να συστήσουμε το Προεδρείο της Επιτροπής μας ε, μέσω της εκλογής του Προέδρου και ε, με τέσσερις αντιπροέδρους. Η σειρά θα έχει ως εξής. Πρώτον θα επιλέξουμε τον Πρόεδρο που τότε θα πάρει τη θέση μου και Έπειτα θα συνεχίσουμε με την εκλογή των αντιπροέδρων. Και έτσι θα ολοκληρωθούν οι σημερινές εργασίες μας μέχρι την επόμενη σύγκληση της Επιτροπής. Θα σας αναγνώσω τα ονόματα των μελών που θα αντικατασταθούν. Η συνάδελφος Κοράτσα Μπίλντ αντικαθίσταται την κυρία Βερέινα, η κυρία Έλβιγκ, συγγνώμη. Ο κύριος Έλβιγκ από τον Ζαγοράκη και ο Περιστούριτς από την Οφίσια Σαϊσέλα. Ο συνάδελφος Μίτσι από τον συνάδελφο Μωρέτη ο συνάδελφος Κραούνλι από τον συνάδελφο Άλαο ο συνάδελφος Σούλικ από τον συνάδελφο Κάλλας και ο συνάδελφος Σόλτερς από τον συνάδελφο Άλμπρεχτ είναι παρόντες ε, οι ανεκαταστάτες. Ε, μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Διαπιστώνω την ύπαρξη απαρτίας που για αυτήν τη συνεδρίαση είναι 10 τουλάχιστον ευρωβουλευτές και αν υπάρχουν συνάδελφοι που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, παρακαλώ ας το πράξουν. Προς το παρόν στο Προεδρείο έχει φτάσει η μοναδική υποψηφιότητα της συναδέλφου Βίκη Φόρντ. Εάν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, ας το πράξουν ευθύς αμέσως. διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει καμία υποψηφιότητα. Υπάρχει μόνο υποψηφιότητα της συναδέλφου Βίκη Φόρντ. La collega, vi propongo che la collega, Ήθελα να σας προτείνω να εκλεγεί διαβοής, αλλά το πράξατε ήδη. Και καλώ την κυρία Φόρντ να έρθει στο Προεδρείο. I've started by remembering my voting card. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στον ορισμό των αντιπροέδρων της Επιτροπής μας. Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ είναι η πρώτη υποψήφια. Από ό,τι κατάλαβα, Μάλλον είχε και αυτή προβλήματα με το Eurostar όπως ε, και άλλοι. Δεν είναι καλή αρχή αυτή σήμερα. Δέχεστε πάντως την υποψηφιότητα. Θέλω πρώτα απ' όλα εκ μέρου ε, τη ομάδα μου να σα συγχαρώ και προσβλέπουμε σε πολύ καλή συνεργασία. Είναι αλήθεια ότι προτείνουμε ε, στη θέση τη πρώτη αντιπροέδρου την κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Δυστυχώ, ναι, έμεινε πολύ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα δυσκολεύεται να έρθει στην υπόλοιπη Ευρώπη Πάντως δέχεται την ε, υποψηφιότητα αυτή και θα δεχτεί τη θέση εφόσον εκλεγεί. Άλλες υποψηφιότητες. Αν ε, δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες, δεχόμαστε τότε την αναμαρια Μαρία Κορατσαμπίλτ και είναι πρόσδεκτη στον Ηνωμένο Βασίλειο όποτε θέλει. Εντάξει, την φανταζόμαστε ότι βρίσκεται εδώ μαζί μα αν και δεν βρίσκεται, αλλά τη φανταζόμαστε. για τη δεύτερη αντιπροεδρία. Ρόμπερτ Ρόσφολτ είναι ο υποψήφιος. Πού είναι, είναι εδώ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα και εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την εκλογή σας. Εκ μέρους της Άλντε θέλω να προτείνω τον Ρομπέρο Σφόρ. Ήταν ιδιαίτερα δραστήριο μέλος της Επιτροπής αυτής την προηγούμενη πενταετία ήταν μάλιστα και συγητής για την προστασία των καταναλωτών. Αν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες, τότε διαβοής εκλέγεται ως δεύτερος αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας, ο κύριος Ροσφόρτ. Ξέρω ότι η κυρία Γκέπχαρτ θα ήθελε να υποβάλει μια υποψηφιότητα για την τρίτη θέση αντιπρόεδρο. σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα εξ από τη σοσιαλιστική ομάδα να σα συγχαρώ, όπω και την κυρία Κοράτσα Μπίλτ και τον κύριο Ροσφόρ, σαν τρίτο αντιπρόεδρο θα ήθελα να προτείνω την κυρία Κάτριν Στάιλερ, η οποία είναι πολύ γνωστή βέβαια συνάδελφος στην Επιτροπή αυτή. can I take it... Μπορώ να θεωρήσω ότι, κυρία, ότι δεν υπάρχουν άλλες ε, προτάσεις για τη θέση του τρίτου αντιπρόεδρου, στην οποία περίπτωση διαβοής ε, εκλέγουμε την Κάτριν Στάιλερ. And the fourth vice Τέταρτη αντιπροεδρία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια Κάθριν. Μια δε, δεύτερη αντιπροεδρία για τους σοσιαλιστές θέλω να προτείνω. Τον αγαπητό μας συνάδελφο Σέζιο Κοφεράτη. Ο οποίος θα μπορεί να επανέλθει λοιπόν στα προεδρικά θεωρία με αυτόν τον τρόπο. Are there any other nominations? Άλλες υποψηφιότητες, στην οποία περίπτωση μπορείτε να ξαναγυρίσετε πάλι σας παρακαλώ, μας λείψατε. Και τώρα να επιβεβαιώσω το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεών μας, το οποίο πιστεύω ότι έχει διανεμηθεί σε όλα τα μέλη προηγουμένως πριν από τη συνεδρίασή μας. Υπάρχουν ε, αντιρρήσεις στο προτινόμενο χρονοδιάγραμμα συναντήσεών μας, συνεδριασεών μας. Όχι, εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι ημερομηνίε αυτές θα είναι οι ημερομηνίε για τη συνεδριάση της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Αυτό ήταν εύκολο. Αυτό ήταν εύκολο. Μπορούμε να, συγχωρήσουμε, να συνεχίσουμε με την ίδια ευκολία. Θα ήθελα απλώ, εάν μου επιτρέπετε, να πω λίγα λόγια και να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για επικείμενες αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε. Ξέρω ότι αυτή η Επιτροπή με την καταπληκτική ηγεσία του προκατόχου μου του Μάλκολμ Χάρμπορ είχε μια πολύ καλή φήμη μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για σκληρή εργασία ώστε να μειωθούν τα φράγμα, οι φραγμοί στην οικονομική ανάπτυξη και για την απλοποίηση της νομοθεσίας ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα σε όλη την εσωτερική αγορά, ενώ συγχρόνως εξασφάλιζε βελτιώσεις υπέρ των καταναλωτών σε πολλούς τομείς πιστεύω και εγώ ότι μια καλά λειτουργούσα ενιαία αγορά μπορεί να απο, απελευθερώσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ευμάρεια στην Ευρώπη προς το όφελος και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Πιστεύω όμως ότι εάν δεν λειτουργήσει σωστά μπορεί να εμποδίσει το επιχειρήν και να οδηγήσει σε μια απολυθωμένη κουλτούρα στι επιχειρήσει. Η ενή αγορά θα πρέπει να βοηθήσει τα άτομα να εκπαιδεύονται σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να πουλούσε πάνω από 500 εκατομμύρια καταναλωτέ. Δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη γραφειοκρατία, η οποία είναι και πολύ δάπανη. Κατά τη δική μου άποψη, η Επιτροπή μα θα πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στι θέσει απασχόληση και τι προτεραιότητε ανάπτυξη και ιδίω στην εφαρμογή και τη σωστή λειτουργία τη υπάρχουσα νομοθεσίας και όχι να επιδιώκει πάντα νέα νομοθετικά μέτρα. Εγώ θέλω να βασιστώ στην φήμη που έχει εδραιώσει η Επιτροπή μας ότι θα είμαστε ανοιχτοί, διάφανοι και θα δίνουμε έμφαση στην ευφυά νομοθεσία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσέγγιση του Malcolm Harbour που αγωνίστηκε με πάθος για να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει πάντα έλεγχος και διερεύνηση για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη διαμόρφωση πολιτικής. Και σας προσκαλώ να χρησιμοποιήσετε την, ε, την, ε, το σύστημα αξιολόγησης του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το οποίο αγωνίστηκε η Επιτροπή μας να γίνει πραγματικότητα. Κατά τη δική μου εμπειρία, αν θέλετε να πετύχετε κάτι σε αυτό το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να έχετε μια καλή σχέση εργασίας και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί υπάρχουν πάντα δύο σκέλη της νομοθετικής εξουσίας και έχουν τονίσει οι ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει η εσωτερική αγορά να βασίζεται περισσότερο στην επικουρικότητα και την αναλογικότητα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το κοινό λοιπόν πλέγμα κανόνων αγοράς δεν σημαίνει ότι θα είναι όλες οι αγορές ταυτόσιμες. Η νομοθεσία όμως των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύπλοκη. Υπάρχει κάτι το θετικό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το δυναμικό της ψηφιακής ενίας αγοράς με το να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτής της αγοράς σε πολλά θέματα και καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Αυτές είναι οι αρχικές μου σκέψεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω που εναποθέτετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα Υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν εργαστεί με την προηγούμενη Επιτροπή και προσβλέπω να συνεργαστώ μαζί σας με τους βουλευτές από όλες τις χώρες και όλες τις πολιτικές ομάδες, με τους συντονιστές, με τους αντιπροέδρους και με όλους εσάς. Και θα ήθελα να ξέρω τις απόψεις σας και τις προτεραιότητες σας σε σχέση με τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει η Επιτροπή μας κατά τη διάρκεια της επικείμενης θητείας σας. Σας ευχαριστώ πολύ και η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή. Και μερικά ακόμα στοιχεία που πρέπει να σας αναφέρω. Την Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα, θα γίνουν ακροάσεις επιτρόπων στο Στρασβούργο για τους επιτρόπους που αντικαθίστανται επειδή εξελέγησαν ως βουλευτές. Η δική μας επιτροπή δεν είναι η κύρια επιτροπή σε σχέση με την αντικατάσταση του κυρίου Ταγιάννη, αλλά ζήτησα τα μέλη της επιτροπής μας να προσκληθούν εφόσον το θέλουν να πάνε στην ακρόαση του αντικαταστάτη του κυρίου Ταγιάννη και φαντάζομαι ότι εάν θέλετε να πάτε σε αυτήν την ακρόαση θα λάβετε μια πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι ανοιχτοί και διάφανοι. Ξέρω ότι η γραμματεία έχουν μια σειρά θεμάτων που θέλουν επίση να συζητήσουν με τους συντονιστές. <clears throat> Προτού κάνουμε τις καλοκαιρινές διακοπές, προτείνουν να γίνει μια συνεδρίαση την επόμενη Πέμπτη ε, πριν από τις ε, ψηφοφορίες του Σασμού Και οι γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν που εμπλέκονται στα θέματα της εσωτερικής αγοράς έχουν προσφερθεί να μας συναντήσουν εγώ θα πρότεινα να υπάρχει μια ανοιχτή συνεδρίαση συντονιστών, ώστε όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να λάβουν μέρο στην ανταλλαγή απόψεων με τι γενικέ διευθύνσει Κομισιόν θα μπορούν να το πράξουν πριν από τι θερινέ διακοπέ και έτσι θα έχετε τον απαραίτητο χρόνο να το κάνετε αυτό. Αυτό θα γίνει το απόγευμα τη 22η Ιουλίου και θα υπάρχει και διερμηνία σε αυτή τη συνεδρίαση. Ένα τελικό σημείο. Κάποιοι θεωρούν ότι θα ήταν ίσως χρήσιμο να έχουμε κάποιες ανταλλαγές απόψεων με τους απερχόμενους επιτρόπους, να ακούσουν ποιες είναι οι απόψεις τους και τα συμπεράσματά τους από την προηγούμενη θητεία. Αυτό ενδεχομένως θα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε στη συνάντηση των συντονιστών, γιατί έχουμε πολλά να διδαχτούμε από την εμπειρία τους και για τον καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα πέντε χρόνια. Εάν ενδιαφέρεστε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια καταληκτική ανταλλαγή απόψεων με κάποιους από τους επιτρόπους οι οποίοι αποσύρονται, μπορούμε ίσως να δώσουμε χρόνο της Επιτροπής μας το Σεπτέμβριο και να το πράξουμε. Νομίζω ότι αυτά ήταν όλα. Σας ευχαριστώ πολύ.